κατευθείαν από την 1η Ιουλίου 2013. Οι αρχές της Πολωνίας μου απίθυναν ένα αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του κ. Μπίκνιεφ Ζιόμπρο και σύμφωνα με το άρθρο 6 πράγραφο 2 του κανονισμού παραπέμπουμε αυτό το αίτημα στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Η συνάδελφος κ. Λάρα Κόμη μου υπέβαλε ένα αίτημα υπεράσπισης της